για την εκπνοή της ε, θητείας τους ως ευρωβουλευτές λόγω του ότι εξελέγησαν στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχεται αυτές τις πληροφορίες και σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του εσωτερικού κανονισμού που αφορά την εκλογή